sitzung wieder aufgenommen. ελπίζω ότι είσαστε αρκετά δυναμωμένοι για την τελευταία ευθεία στην οποία βρισκόμαστε, την τελική ευθεία. Εφέτος ε, τα πρακτικά έχουν διανεμηθεί, εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, θεωρούνται ότι έχουν εγκριθεί. Ακολουθεί η συζήτηση για θέματα δημοκρατίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμάτων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για μία ώρα και ξεκινάμε την κατάσταση στη Δημοκρατική Δημοκρατία του Κόγκο. Δίνω το λόγο στην κυρία Γκάμπριελ καταρχήν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κρίση στην επαρχία Κιβού ε, ανέδειξε παλιές ε, ε, εντάσεις και προβλήματα πολύ σοβαρά που δυστυχώς η κογκολέζικη κυβέρνηση δεν τα είχε αντιμετωπίσει. Η ατιμορρησία και η έλλειψη επαγγελματικού στρατού, ε, ο ανταγωνισμός για τον έλεγχο των φυσικών πόρων δείχνει την έλλειψη της πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης να προβεί σε μεταρρυθμίσεις. Έτσι, το βάρος της ανασφάλειας που πλήττει τον πληθυσμό του Κογκό είναι δυσβάσταχτο πια. Θα πρέπει επιτέλους να κάνουμε κάτι για να επιληθεί αυτή η σύγκρουση και να μην αρκούμαστε σε απλή διαχείρισή της. Και γι' αυτό τρεις ε, είναι οι λέξεις κλειδιά, διάλογος, ε, υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα. Ε, ευθύνη, υπευθυνότητα, πρώτα απ' όλα κογκολέζικη, κοινωνική, οικονομική, ε, πολιτική, άμεση κατάπαυση των βιοπραγιών, συνεργασία με το Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο, λειτουργική απονομή τη δικαιοσύνη και ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλε αυτέ είναι οι προποθέσει που θα μα επιτρέψουν να ξεπεράσουμε την κρίση και όχι να περιοριστούμε σε απλή διαχείριση. Σε περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει ο διάλογο μεταξύ Ρουάντα, Ουγγάντα και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό να συνεχιστεί. Έχω ένα επιπλέον λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να το αξιοποιήσω, αν γίνεται. Εγώ έχω μονάχα ένα λεπτό στη διάθεσή σας, σύμφωνα με τον κατάλογο, λέει ο πρόεδρος Βίλαντ. Σας παρακαλώ όμως να μιλάτε και πιο αργά, διότι δεν, προ... σας προφταίνουν τα μηχανήματα διερμηνίας. Καλώς. Θα συνεχίσω λοιπόν με το περιφερειακό επίπεδο. Θα πρέπει ο διάλογο που έχει ξεκινήσει μεταξύ Κονγκό, Ρουάντα και Ουγγάντα να συνεχιστεί και οι δράσει ε, τη διάσκεψη για την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών και τη Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχιστούν για να καταλήξουν σε βιώσιμη λύση. Θα πρέπει να θεσπιστεί ένα μηχανισμό ε, κοινού ελέγχου με ε, ακατάλληλους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους και τέλος τα ενδιαφερόμενα κράτη από την έκθεση του ΙΕ θα πρέπει να δώσουν κάποιες απαντήσεις στα ερωτήματα που τίθενται στην έκθεση και τέλος σε διεθνέ επίπεδο η Μονούσκο θα πρέπει να υλοποιήσει καλύτερα την αποστολή τη σταθεροποίηση. Αυτό περιμένει ο πληθυσμό και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει ε, σημαντική ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά έχουμε και δύο βασικέ αποστολές, USEC και UPOL. Θα συνεχίσουμε τι προσπάθειε. Και τέλο, μία έκκληση προ την κοκολέζικη κυβέρνηση να κάνει ό,τι μπορεί για να εξασφαλίσει την προστασία του δόκτωρα Μουτβέγκε μετά την απόπειρα δολοφονία του. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για τη ζωή του δόκτωρα Μουτβέγκε, αλλά μιλάμε για όλε αυτέ τι γυναίκε που είναι θύματα σεξουαλική βία ε, και θα έπρεπε να τι προστατεύσει η κογκολέζικη κυβέρνηση. Περιμένουμε μια πολιτική χειρονομία και ένα πολιτικό ε, διάβημα από την κογκολέζικη κυβέρνηση. Ελπίζουμε να τα πράξει. Εγώ κατάλαβα ότι υπάρχει ένα σφάλμα από τις υπηρεσίες. Είχατε πράγματι δύο λεπτά, αλλά παρακαλώ να, να ζητήσω... Στα του να παραμείνετε στα πλαίσια του φυσιολογικού σας χρόνου εργασίας. Αλλιώς... Ε, ε, θα ξεπεράσουμε το χρόνο μας και ε, παρακαλώ ο καθένας να μιλά με κανονικό ρυθμό και να μην ε, μιλά πολύ γρήγορα γιατί αν δεν σας προλάβουν οι δερμήνες θα περάσει και το μήνυμά σας. Κυρία Κρέτσου, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. θα ήθελα να πω ότι ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα με την επαρχία του Βόρειου Κιβού και με την εισβολή του αντάρτητου κινήματος ΜΗ23 στην πόλη της Γκόμα. Δεν μιλούμε απλώς για εμφύλιο πόλεμο στη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Έχουμε έναν άγριο πόλεμο με συμμετοχή πολλών χωρών, η χειρότερη ε, σύγκρουση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γίνεται πόλεμος για τον έλεγχο του ορυκτού πλούτου. Και έχουμε χιλιάδες ε, Πρόσφυγε από την κόμμα. Τα παιδιά δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο, αλλά στρατολογούνται υποχρεωτικά στο στρατό. Έχουμε μαζικές εκτελέσεις, μαζικούς βιασμού. εκφοβισμό του πληθυσμού. Θα πρέπει να γίνει κατεπηγόντω μια επαναξιολόγηση της αποστολή διαφύλαξης της ειρήνης. Δεν νομίζω ότι οι 2.000 ε, κιανόκρανοι και τα ντρόμς που έχουμε εκεί αρκούν για να ελέγξουν την κατάσταση. Ο άμαχος πληθυσμός μένει ανήμπορος και απροστάτευτος. Χρειαζόμαστε μια νέα στρατηγική για να καταπολεμήσουμε την ανταρσία και να προστατεύσουμε τον άμαχο πληθυσμό. Επίσης, να ελέγξουμε και τα κέρδη από τις παράνομες εξορρυκτικές δραστηριότητες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κρέτου. Για δύο λεπτά κύριος Κίλνιλσον. Merci, Président Κυρία Κίλνιτσα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στη δημοκρατική δημοκρατία του Κονγκό υπάρχει μια λέξη η οποία συνοψίζει την κατάσταση αυτής της περιοχής. Μακαλά. Είναι ένα χρυσορυχείο στο βόρειο τμήμα του Κονγκό που είναι συμβολικό της ε, λαιλασία που λαμβάνει η χώρα στι μεγάλες λίμνες, στην περιοχή των μεγάλων λιμνών και στο Κονγκό. Υπάρχει η δράση λοιπόν των πολιτοφυλακών και των, ε, φυλά... Ε, πολεμάρχων οι οποίοι θέλουν να διώξουν τους εργαζόμενους από εκεί και είναι και ένας χώρος απόλυτης ατιμορρησίας. Η κυβέρνηση του Κονγκό είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη. Η... Τα συμφωνιστικά ιδρύματα δεν έχουν καμία απολύτως παρουσία ζητούν από τους κρατούμενους να δώσουν εγγυήσεις για να συνεχίσουν εκεί. Είναι ένας χώρος όπου πεθαίνει ο κόσμος. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα διατροφής. Υπάρχει υπερπληθυσμός, γίνονται βασανιστήρια για όλους αυτούς που είναι εκεί. Το Μάκαλα είναι το σύμβολο της περιοχής αυτής στο Κονγκό. Μία ειρήνη στο Κονγκό προϋποθέτει την επαναφορά του κράτους δικαίου και της δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να γίνει η ειρήνη σε βάρο τη δικαιοσύνη. Πρέπει να είμαστε σαφεί. Οποιαδήποτε συμφωνία ειρήνη θα πρέπει να ε, μην περιλαμβάνει οποιαδήποτε μορφή ατιμορρησία για όλου αυτού οι οποίοι έχουν ελεηλατήσει και επιπολίσει αυτή τη χώρα. Το να αγωνιστούμε κατά της ατιμορρησία στη χώρα αυτή, όπου πάνω από 2 εκατομμύρια γυναικών έχουν σκοτωθεί τα τελευταία 6 χρόνια, αυτό πρέπει να κάνει ο Δόκτωρ Μουντβέγκε, ο υπερασπιστή των βιασμένων γυναικών παρά τι βιαιότητε και τι ακρότητε, εξακολουθεί να κάνει ένα τεράστιο έργο για τι γυναίκε και γι' αυτό προσπαθήσαν να τον δολοφονήσουν. Αυτέ οι πράξει πρέπει να καταδικαστούν, αλλά κυρίω να ασκήσουμε πίεση στην κυβέρνηση του Κονγκό, ώστε αυτή η απόπειρα δολοφονία να αποτελέσει αντικείμενο δικαστική έρευνα στο του δυνατό. Η ειρήνη περνάει και από τη μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη, δηλαδή να υπάρξει σωστή διανομή των φυσικών πόρων του Κονγκό. Σας ευχαριστώ κύριε Κίλνιτσεν για ένα μισή λεπτό η κυρία Ογιούλαντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Οι συγκρούσεις που έχουν οδηγήσει στο θάνατο χιλιάδων ανθρώπων στο Κονγκό έχουν κάνει την δημοκρατική δημοκρατία του Κονγκό σε μια εμπόλεμη ζώνη όπου οι πολέμαρχοι και οι διεφθαρμένοι αξιωματούχοι είναι οι μόνοι οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση. Δυστυχώ η διεθνή κοινότητα δεν έχει δώσει την απαραίτητη υποστήριξη και τα απαραίτητα αποτελέσματα η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ υπάρχει επιτόπου για 13 χρόνια, κάθε χρόνο κοστίζει 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Παρ' όλα αυτά δεν υπήρξε κάποιο αποτέλεσμα. Η κίνηση M23 εξακολουθεί να έχει την εξουσία στην ανατολική περιοχή του Κονγκό και δεν θα είναι η τελευταία τέτοια κίνηση η οποία ελέγχει οι περιοχές του Κονγκό. Χρειαζόμαστε μια ε, πραγματικά οραματιστική και δυναμική στάση για να υπάρξουν πολιτικοί θεσμοί στο Κονγκό οι οποίοι θα εγγυηθούν τα θεμελιώδη δικαιώματα. Μέχρι στιγμής δυστυχώς δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ κυρία Ογιουλάντ. Από τους συντάκτες του ψηφίσματος λαμβάνει το λόγο στο τελευταίο ο κύριος Μέρφυ για δύο λεπτά. Η πρόσφατη κλιμάκωση της βίας στις ανατολικές επαρχίες του Κονγκό μετά από την εξέγευση τμήματων του στρατού και την είσοδο στην κόμμα ανταρτών είναι μια πάρα πολύ κρίση, πολύ μεγάλη κρίση που διαδέχεται μια εξίσου μεγάλη κρίση και πάει λέγοντας. Υπάρχουν διάφοροι πολέμαρχοι στην περιοχή οι οποίοι εδώ και δεκαετίες προσπαθούν να καταπολεμήσουν τα αντιτιθέμενα συμφέροντα και να εκμεταλλευτούν τα συμφέροντα τα οικονομικά της περιοχής. Όλες οι ομάδες οι αντάρτικες μαζί και ο στρατός έχουν παραβιάσει μαζικά με τρομοκρατικό τρόπο τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχουν ασκήσει ακόμα και σεξουαλική βία. Κάθε ώρα βιάζονται 50 γυναίκες, 48 γυναίκες ε, στην χώρα και 4,5 εκατομμύρια ε, κάτοικοι της περιοχής έχουν χάσει τη ζωή τους από το 1998 και μετά. Και ε, λόγω των τελευταίων συγκρούσεων 140.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να αυτοεκτοπιστούν ουσιαστικά Έχει υπάρξει βέβαια μια προσπάθεια για αποκατάσταση της ε, σταθερότητας στην περιοχή μέσω 20.000 ε, στρατιωτών των Ηνωμένων Εθνών έτσι ώστε να διασφαλιστεί η λαιλασία αλλά με τακτικό τρόπο των οικονομικών πόρων και των φυσικών πηγών της περιοχής. Είναι πολύ πλούσια η περιοχή αυτή λόγω των φυσικών πόρων οι πολέμαρχοι και οι επίσημοι της κυβέρνησης γίνονται εκατομμυριούχοι μέσω των αμοιβών από τις πολιεθνικές οι οποίες ελέγχουν τους φυσικούς πόρους. Συνεχίζεται ουσιαστικά η απικιοκρατική και υπεριαλιστική επίθεση η οποία έχει γδίσει πλέον τον κόσμο από τους φυσικούς, τις φυσικούς του πόρους αυτός ο κύκλος ο φρικτός της πρέπει να σταματήσει, πρέπει να σταματήσει πια. Είναι απαραίτητο οι φυσικοί πόροι να βρίσκονται στα χέρια της δημοκρατικής εξουσίας και να ωφελούν το σύνολο του πληθυσμού. Ευχαριστώ κύριε Μέρφη. Εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων, ο κύριος Πόσελ καταρχήν για ένα λεπτό το Κίβου και το Κονγκό εν γέννη, παρά το παραδείσιο του οποίο είναι μία από τις πιο ερημωμένες περιοχές του κόσμου. Ενώ θα μπορούσε να είναι παράδεισος πάνω στη γη, είναι μία κόλαση. Είναι μια από τις πλουσιότερες δυνητικά χώρες της Αφρικής το Κονγκό. Θα μπορούσε με τους υδάτινους πόρους να τροφοδοτεί όλη την Αφρική. Θα μπορούσε να ήταν ένα κέντρο παραγωγής τροφίμων για όλη την Αφρική. Έχει τεράστιες πηγές πρώτων υλών και θα μπορούσε να έχει μια τεράστια βιομηχανία. Αλλά λόγω της ιστορίας του, της απικιακής και της μεταπικιακής είναι έρμεο πολέμων και διεφθαρμένων κυβερνήσεων. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν ό,τι είναι δυνατόν τεστ αυτή η κεντρική περιοχή της Αφρικής να περάσει σε μια κατάσταση ειρήνευσης. Αυτό γίνεται μονάχα μέσα από μια στενή συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρικανική Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη. Οι συμφωνίες οι οποίες γίνονται σε διμερές επίπεδο όπως αυτή των μεγάλων λιμνών χωρίς να εφαρμοστούν στην πράξη είναι μια καταστροφή για την περιοχή αυτή. Εμείς θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στην κυβέρνηση του Κονγκό να έχει μια διάρκεια στον χρόνο. Ευχαριστώ κύριε Πόσελτ. Για 1,5 λεπτό έχει το λόγο η κυρία Γκούρμαϊ. Κύριε η ένοπλη εξέγερση μεταξύ ε, επίσημου στρατού και μη 23 έχει οξύνει την κατάσταση και έχει επαναφέρει συγκρούσεις. Η κατάσταση παρά τα ψηφίσματά μας εξακολουθεί να είναι σταθερή. Είναι πολλά τα αίτια αυτής της σύγκρουσης και πολλές συνέπειες της όλη την περιοχή. Γι' αυτό και θα πρέπει κατεβηγόντως να αναλυφθεί μια στρατηγική. Παρά την ε, εθνική κατάσταση, το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, ε, η ανάμειξη των γειτονικών χωρών και το θέμα της εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη γιατί οι παράνομες δραστηριότητες ε, εξορυκτικές ε, θα πρέπει να παρεμποδιστούν μέχρι ότου βρεθεί οριστική λύση. Επαναλαμβάνω, είναι τεράστιες φρικαλαιότητες που έχουν υποστεί ε, οι πολίτες του Κονγκό με μια κατάσταση που έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερα χρήση σεξουαλικής βίας σε, μαζικούς, σε μαζικές διαστάσεις κατά νεαρών κοριτσιών και γυναικών. Είναι αποτρόπαια τα εγκλήματα αυτά. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τα θύματα να ανακάμψουν κάμψουν και ψυχολογικά και σωματικά. Είναι τεράστιες οι συνέπειε τη σύγκρουση αυτή και πρέπει να αντιμετωπιστούν σοβαρά. Χωρί σωστή στρατηγική για δημο... επαναδημοκρατισμό και επαναφορά των... αποστρατικοποίηση και επαναφορά των στρατιωτών στην κοινωνία, δεν θα μπορέσουμε να βρούμε μακροχρόνια λύση. 1,5 λεπτό κύριε Σάκε. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ένα τοξικό μείγμα βία πάνω από του φυσικού πόρου, βία, βιασμοί, στρατολόγηση παιδιών, όλα αυτά αποσταθεροποιούν το Κονγκό και αφορούν μια κοινότητα πάνω από 2,5 εκατομμύρια ανθρώπων. Οι στρατιωτικέ ομάδε και οι παραστρατιωτικέ ομάδε κάνουν τα χειρότερα εγκλήματα με τη βοήθεια των γειτόνων του Κονγκό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δράσει με έναν τρόπο που ήταν συντονισμένο μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη και την Αφρικανική Ένωση για να υπάρξει ένα τέρμα σε αυτή την πολεμική κατάσταση και επίσης για να εμποδίσει μια περαιτέρω επέκταση στην ευρύτερη περιφέρεια των μεγάλων λιμνών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δράσει στεναρά και από κοινού. Υπάρχουν ορισμένα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν διακόψει τη βοήθεια προς τη Ρουάντα λόγω της έκθεσης του ΟΗΕ που δείχνει ότι η Ρουάντα είναι με πλεγμένη στους Στι συγκρούσει στο Κονγκό. Χρειαζόμαστε επίση και μια κοινή θέση εναντίον όλων αυτών που έχουν παραβιάσει το εμπάργο όπλων του Ηνωμένου του ΟΗΕ. Μπορούμε να κάνουμε και περισσότερα με το να βελτιώσουμε τη διαφάνεια σε σχέση με τα ορυκτά τα οποία εξορίσσονται παρανόμω. χρειαζόνται περισσότερε λοιπόν έρευνε για τα θέματα αυτά. Αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει εγκρέματα, πολέμου εγκρήματα κατά της ανθρωπότητας, σεξουαλική βία κατά των γυναικών και έχουν ε, στρατολογήσει παιδιά στρατιώτε. όλοι αυτοί πρέπει να έρθουν ενώπιον τη δικαιοσύνης. Θα πρέπει να σταματήσει η ατιμορρησία και θέλω να δώσω ιδιαίτερη έμφαση στην επίθεση κατά του θαραλέου δόκτωρα Μουγκέβιου που οδήγησε στο θάνατο του σωματοφύλακά του. Όλα αυτά πρέπει να τύχουν ανεξάρτητη έρευνα. Έχει βοηθήσει πάρα πολλέ γυναίκε που είναι τα κύρια θύματα τη συνεχιζόμενη βία στο Κόγκο. Σα ευχαριστώ κύριε Σάκε. Ο κύριο Πάσκα για ένα μισή λεπτό επίσης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι οι συνεχιζόμενες βιοπραγίες στην ανατολική περιοχή της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό είναι απόρρια του πολέμου και των συγκρούσεων για τον έλεγχο του ορυκτού πλούτου. Ε, οι αντάρτες κάνουν ό,τι μπορούν για να εκμεταλλευτούν την κατάσταση και οι γειτονικέ χώρες υποδαβλίζουν αυτή τη σύγκρουση για να έχουν πρόσβαση στον ορεικτό πλούτο. Και μάλιστα ο πληθυσμός έχει γίνει θύμα των εξορρυκτικών βιομηχανιών και με τη βοήθεια ένοπλων παραστρατικών δυνάμεων εκμεταλλεύεται τον ορεικτό πλούτο του Κονγκό. Αυτό που κάνουμε συνήθως είναι να σταθεροποιήσουμε, να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να σταθεροποιήσουμε την πολιτική κατάσταση στη χώρα. Στην περίπτωση όμως της λαϊκής δημοκρατίας του Κονγκό θα πρέπει πρώτα απ' όλα να σταματήσουμε τις εμπορικές συναλλαγές ε, και τη παράνομη εξορρυκτική δραστηριότητα. Με βάση το νόμο Dodd-Frank του Αμερικανικού Κογκρέσου θα μπορούσαμε να επιβάλλουμε και εμείς συχνηλασιμότητα των προϊόντων αυτής της εξορρυκτικής δραστηριότητας για να αποφύγουμε την αγοραπολισία παράνομων ορυκτών στην παγκόσμια αγορά. Μια τέτοια χνηλασιμότητα των ορυκτών ίσως σταματήσει τις εθνικές συγκρούσεις γιατί δεν θα είναι πια το κέρδος ε, κίνητρο για την ε, συνέχιση του. Σας ευχαριστώ. Οι υπόλοιποι ομιλητές, ο κύριος Πέντα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αν έχω κάνει σωστή καταμέτρηση, είναι η έκτη φορά μέσα στην τρέχουσα νομοθετική περίοδο που συζητούμε για την τόσο δύσκολη κατάσταση στη δημοκρατική δημοκρατία του Κονγκό. Έχουμε αντιμετωπίσει ήδη τα θέματα αυτά και έχουμε τώρα ένα ψήφισμα ενώπιόν μας και επίσης και η Ισομερή Συνέλευση ΑΚΕ ε, ΕΟΚ η οποία, ήταν στο, η οποία έλαβε χώρα στο Σουρινάμ πρόσφατα, κατέληξε και αυτή σε μια κοινή δήλωση. Πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερο συντονισμό με τα Ηνωμένα Έθνη και με του περιφερειακού εταίρου. Αυτό το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε την εφαρμογή αυτού του κοινού ψηφίσματο σε συνεργασία και με τις, τους διάφορους διεθνούς φόρους. Ευχαριστώ κυρία Πρέντα. Ο κύριος Ρέπο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε ειδήσει για την βία που σοβεί στο Ανατολικό Κονγκό και είναι ανησυχητικά όλα αυτά τα στοιχεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την ε, ασφάλεια όλων αυτών των ανθρώπων στην περιοχή και επίσης να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση για τις ανθρωπιστικές οργανώσεις. Η Αφρικανική Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ΟΗΕ έχουν, να διαδραματίσουν όλοι ένα ρόλο από κοινού μέσα στην δημοκρατική δημοκρατία του Κονγκό. Έχουμε ασύλληπτες μορφές βίας, μαζικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μαζικούς βιασμούς, που χρησιμοποιούνται ως όπλο πολέμου. Υπάρχουν λοιπόν μαζικές παραβιάσεις οι οποίες θα πρέπει να έλθουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Εάν δεν υπάρξει ε, τιμωρία, τότε θα συνεχιστεί αυτό το κλίμα της ατιμορρησίας που θα οδηγήσει σε περαιτέρω βία. Ευχαριστώ κύριε Ρέπο. Ερχόμαστε στη διαδικασία οφθαλμοσυλληπτικού χαρακτήρα και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Κορχολά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κατάσταση στην ανατολική αυτή περιοχή του Κογκό είναι πραγματικά καταστροφική. Εδώ και 7 μήνες η ομάδα M23 λαιλατεί συστηματικά παραβιάζονται με σοβαρό τρόπο τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπάρχουν μαζικοί βιασμοί γυναικών και παιδιών, βασανιστήρια και χρήση ε, παιδιών στρατιωτών. Η δε ανθρωπιστική κρίση βαθαίνει συνεχώς. Υπάρχει ένα μεγάλο αίσθημα ατιμορρησίας γιατί αυτά τα εγκλήματα πολέμου δεν διώκονται. Και οι τεράστιοι φυσικοί πόροι του Ανατολικού Κογό χρησιμοποιούνται από τους λάθος ανθρώπους και ωφελούν τις ένοπλες ομάδες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη θα πρέπει επιτέλους κάτι να κάνουν για να λυθεί το πρόβλημα και να σταματήσει αυτή η ανθρωπιστική καταστροφή. Οι ένοχοι βασανιστήριων και βιασμών πρέπει να τιμωρηθούν. Σας ευχαριστώ κύριε Κόρχορε. Ο κύριος Κούκαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με ανησυχεί ιδιαίτερα η ανθρωπιστική κρίση. Έχουμε μαζικές καταπατήσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Θα πρέπει να καταδικάσουμε τους μαζικούς βιασμούς, τα βασανιστήρια, σφαγίες πολιτών και στρατολόγηση παιδιών στρατιωτών. Η μη προσαγωγή των αυτούργων καταστρατήγη ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενισχύει το αίσθημα της ατιμορρησίας και ενθαρρύνει την περαιτέρω διάπραξη αξιόπινων ενεργειών. Και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει εδώ. Θα πρέπει να συμβάλλουμε στην αποκατάσταση της δικαιοσύνης και της ασφάλειας στη χώρα και να εξασφαλίσουμε τη συνέχιση της αποστολής USM και UPOL. Είναι σημαντικό να βρούμε μια λύση που θα εξασφαλίζει το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα επαναφέρει ασφάλεια, ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ακολουθεί κύριε Γκέρνια το Ευχαριστώ. Η ανταρσία του M23 κατά του στρατού διατάραξε το σύστημα της ασφάλειας και το οδήγησε τεράστιες ε, απώλειες στο λαό. Ε, το M23 ε, προσπάθησε να αντιταχθεί στον ένα στρατό με αποτέλεσμα να έχουμε δύο εκατομμύρια πρόσφυγες και χιλιάδες που, που έτρεξαν προς την Ρουάντα ή την Ουγγάντα. Έχουμε μαζικούς βιασμούς και βασανιστήρια τεράστια ανησυχία δημιουργείται στην παγκόσμια κοινότητα εξαιτία τη κοινωνική, οικονομική και πολιτική κρίση στο Κονγκό. Θα πρέπει να καταδικάσουμε οποιαδήποτε βιοπραγία και καταστρατήγηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να τιμωρηθούν ε, αυστηρά όσοι ε, διέπραξαν εγκλήματα. Η λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό θα πρέπει να επανέλθει σε σταθερότητα και δημοκρατία με ανεξάρτητους θεσμούς με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας με πιο συντονισμένο και αποτελεσματικό τρόπο ε, προκειμένου να εξασφαλίσουμε η ιατροφαρμακευτική και ανθρωπιστική περίθαλψη σε όλα τα θύματα της συγκεκριμένης σύγκρουσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Γκέρνγκερ. Εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να σας... Ε, ε, έχω μονάχα τα, τις απελπισμένες εκκλήσεις των διερμηνέων όταν μιλάτε τόσο γρήγορα. Κύριο Σκέλη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι τραγική η κατάσταση στο Κονγκό αν σκεφτείτε ιδιαίτερα ότι αυτή η χώρα θα πρέπει να, θα πρέπει να ήταν μια από τις πλουσιότερες στον χώρο, στον κόσμο, λόγω των φυσικών πόρων της, αλλά δεν συμβαίνει αυτό. Όπως έχει ήδη ακουστεί, αν και η δημοκρατία του Κονγκό είναι ανεξάρτητη εδώ και μισό αιώνα, δεν έχει υπάρξει πραγματική πρόοδος για την αποκατάσταση της δημοκρατίας και τον σεβασμό του κράτους δικαίου. Σαν συνέπεια λοιπόν, η τυφλή βία συνεχίζεται, επεκτείνεται και μάλιστα πρόσφατα είδαμε ότι λαιλατήθηκαν ανάμεσα σε άλλα 600 σχολεία. Δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος με τον τρόπο αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να σταθεροποιήσουμε τη χώρα και δεύτερον θα πρέπει χώρες όπως η Ουγγάντα και η Ρουάντα να αποχωρήσουν, να μην παρεμβαίνουν για να μπορέσουν να βοηθήσουν αυτοί οι οποίοι έχουν την πραγματική διάθεση. Ευχαριστώ κύριε Κέλλη. Ο κύριος Λίζεκ. Ευχαριστώ. Φυσικά η πολιτική κατάσταση στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και η ανθρωπιστική κατάσταση είναι δραματική. Βέβαια δεν θα επιλύσουμε τα προβλήματα αυτά αν δεν ε, αποκλιμακώσουμε την κρίση ιδιαίτερα μεταξύ του Κονγκό και της Ρουάντας. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να ασκήσουμε πιέσεις ώστε οι κυβερνήσεις των γειτονικών χωρών να μην στηρίζουν, να συνεχίσουν να στηρίζουν τους αντάρτες ε, και να μην έχουμε διακρίσεις λόγω συμμετοχής σε θρησκευτικές ή πολιτικές μειονότητες. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την διαπραγμάτευση μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών και να αποκλιμακώσουμε την ένταση κυρίως στην ανατολική πλευρά του Κονγκό να ενισχύσουμε την Μονούσκο και να ε, παρεμποδίσουμε την παράνομη εξόριξη δραστηριοτήτων. Σημαντικό είναι να επαναφέρουμε ένα μηχανισμό πιστοποίησης ε, των ορυκτών προϊόντων από την περιοχή του Κίμπερλε. Για να κλείσουμε τη συζήτηση, είναι το λόγο στον Επίτροπο κ. Τσόλο. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, έντιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χαιρετίζουμε την ε, πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να ψήσουμε σε σχέση με τη Δημοκρατική Δημοκρατία του Κονγκό και ιδίω για την κατάσταση στο Ανατολικό Κονγκό. Αυτή η κατάσταση ανησυχεί την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχει δώσει δηλαδή στην ε, υιοθέτηση πολλών δηλώσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και, και στα συμπεράσματα επίση έχει αναφερθεί σε δύο από τα τελευταία Συμβούλια Υπουργών Εξωτερικών. Συμμεριζόμαστε τι ανησυχίε που αναφέρονται στο κατεπήγον ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είτε σε ό,τι πρόκειται για την ανθρωπιστική κατάσταση, την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδίω τη σεξουαλική βία και τη ανάγκη να σταματήσει η δράση των ενόπλων πολιτεοφυλακών και να επαναέλθει το κράτο δικαίου και η ευκυβερνησία στο ανατολικό τμήμα τη χώρα, κάτι το οποίο περιλαμβάνει και τη μεταρρύθμιση στον τομέα της ασφάλειας και τον αγώνα κατά της παράνομης εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων. Στα πλαίσια αυτά, η κυριαρχικότητα και η εδαφική ακεραιότητα της δημοκρατικής δημοκρατίας του Κονγκό ήταν πάντα μία αρχή επί της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να δεχτεί καμία, κανένα συμβιβασμό. Και έχουμε χωρίς καμία περιστροφή καταδικάσει τις δράσεις των ένοπλων ομάδων στην, ε, στην, στο Ανατολικό Κονγκό και ιδίως της ομάδος ΜΗ-23. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τονίσει ότι είναι απαράδεκτο να δοθεί εξωτερική βοήθεια στην ΜΗ-23 και έχουμε επίσης κάνει μια έκκληση να σταματήσει η ατιμορρησία και να έλθουν ενώπιον των δικαστηρίων όλοι οι ένοχοι εγκληματικών πράξεων. Θεωρούμε επίσης ότι ο καθένας θα πρέπει να καταβάλει συγκεκριμένε και επικοδομητικέ προσπάθειες ώστε να εξευλεθεί μια μόνιμη λύση στην κρίση αυτή. Αυτό απαιτεί τη δημιουργία πολιτικής συνένεση μεταξύ των πολιτών του Κίβου που είναι τα πρώτα θύματα της κρίσης αλλά επίσης και μεταξύ της Δημοκρατικής δημοκρατία του Κόγκο και των γειτόνων τη. ώστε να επιτευθεί μια θετική δυναμική σε περιφερειακό τοπικό επίπεδο που να εξασφαλίσει την ειρήνη, την ασφάλεια και την ανάπτυξη στις μεγάλες λίμνες. Χρειάζεται επίσης να υποστηρίξουμε και το διάλογο μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών στην σύραξη αυτή και επίσης και τις επαφές μεταξύ του Προέδρου της ε, Δημοκρατίας του Κονγκό και της Ρουάντα, της Ουγγάντα σε σχέση με την ειρήνευση στην περιοχή των μεγάλων λιμνών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή και αυτή επίση έτοιμη να δώσει την πολιτική τη συνεισφορά σε πρωτοβουλίε αυτού του είδου για να μπορέσει να υπάρξει μια μόνιμη λύση στην κρίση τη περιοχή. Λαμβάνοντα υπόψη βέβαια την πολυπλοκότητα τη κατάσταση, ζητά μια συνεργασία και μια συμπληρωματικότητα σε ό,τι αφορά τις ενέργειές της και έναντι των ε, εξωτερικών φορέων όπως είναι η η Ένωση για την Ανάπτυξη τη Μεσημερινής Αφρικής, η Επιτροπή για την Αντιμετώπιση των Προβλημάτων στι Μεγάλες λίμνε και επίσης οι οργανώσει του ΟΗΕ στην Δημοκρατική Δημοκρατία του Κονγκό. Και εν σχέση με όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκφράσει κάτι επανάληψη μια θετική γνώμη σε σχέση με τον διορισμό ενό ειδικού εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να συμβάλλει στην επίτευξη μια μόνιμη ειρήνευση στην περιοχή. Θέλω επίση να σα αναφέρω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει όλου του φορεί τη κοινωνία των πολιτών που δρούν καθημερινά υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ενθαρρύνουν το διάλογο μεταξύ, το διάλογο μεταξύ των ακτιβιστών και τη κυβέρνηση. Πάνω από 30 σχέδια αυτή τη στιγμή είναι υποχρηματοδότηση στα πλαίσια των διαφορών θεματικών γραμμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση για συνολικό ποσό άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Σα πληροφορώ επίση ότι Επίτροπος Πίμπαλτς είναι έτοιμος να ξεκινήσει μια ειδική πρωτοβουλία η οποία συνδέεται με την προβληματική της βίας που οφείλεται στο, στο φύλλο. Θέλει να τονίσει την ανάγκη επαναβάθμισης του ρόλου των γυναικών σε εθνικό επίπεδο. Με τα 27 εκατομμύρια ευρώ θα υπάρξουν σχέδια στο πλαίσιο αυτό με την συμμετοχή και άλλων εταίρων όπως είναι τα κράτη-μέλη ώστε να υπάρξει μια ευρύτερη δράση στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Πίτροπε και Έχουμε 7 ψηφίσματα τα οποία έχουν κατατεθεί και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αμέσως μετά τη